Good afternoon to everybody present here in the room or at home or... Uh, Καλησπέρα σε όλους σας, όλοι είσαστε εδώ στο σπίτι. Είμαστε γύρω-γύρω. Καλημέρα. Ξεκινάμε τη συνεδρίαση των προϋπολογισμών και πρώτα απ' όλα μερίσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεύτερο σημείο. Ανακοινώσεις του Προέδρου Τις αποφάσεις των συντονιστών μπορείτε να τις βρείτε στους φακέλους σας. Και αν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση, θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στις ανακοινώσεις. Ωραία. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οπότε σας παρακαλώ πάρα πολύ προσεκτικά να, ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας έχουμε στείλει και να έρθετε σε επαφή με τη γραμματεία εφόσον αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με την ε, διαδικασία. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει σήμερα. 15 και 45 με 5 η ώρα σήμερα το απόγευμα. Η δεύτερη ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 28 του μηνός από τις 16 και 45 μέχρι της 18, 6 ώρα δηλαδή. Υπάρχει διερμηνία στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα αγγλικά, στα ελληνικά, στα πολωνικά και τα πορτογαλικά. Τρίτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε την έγκριση των πρακτικών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα της 17ης και 18ης Φεβρουαρίου. Ε, θα ψηφίσουμε, αλλά πριν ψηφίσουμε θα ήθελα, παρακαλώ, όπως έχουμε προβλέψει και άλλες φορές, θα ζητήσω από τους συζητητές και μόνο από τους συζητητές παρακαλώ να μας παρουσιάσουν το σχέδιο έκθεσής τους. Και σας παρακαλώ επίσης να προσπαθήσετε να τηρήσετε και τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Οπότε το πρώτο σημείο είναι το σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη και έχει να κάνει με τον προπολογισμό το 2021, τμήμα 3. Ο κύριος Λαρουτούρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, όπου και αν βρίσκεστε εδώ ή στις χώρες σας. Η κυρία Φοντελάιν μόλις μας παρουσίασε τις προτάσεις της για την ανάκαμψη της οικονομίας από του χρόνου. Ο προπολογισμό του 2021 λοιπόν ε, θα πρέπει να αποτελέσει και το πρώτο έτος του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου και γι' αυτό έχει τεράστια σημασία για όλους μας, το γνωρίζουμε. Σε δύο μήνες, εκατομμύρια από τους συμπολίτε μας, βρέθηκαν στην ανεργία και δεν ξέρουμε τα επόμενα χρόνια πώς θα ανακάμψει η οικονομία. Έχουμε την κοινωνική κρίση, τη υγεία, την οικονομική, κοινωνική. Πρέπει να κάνουμε κάτι αν θέλουμε να αποφύγουμε το χάος και αν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κερδίσει σε νομιμότητα διότι θα πρέπει οι απαντήσεις να ξεπερνούν τα εθνικά πλαίσια. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ενισχυτικό πλαίσιο, με χαρά σας ανακοινώνω σήμερα ότι αποφασίσαμε να συμφωνήσουμε έξι πολιτικές ομάδες με διαπραγματεύσεις για μήνες. Καταφέραμε λοιπόν να καταλήξουμε σε συμφωνία. Οι έξι αυτές πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ τον Κάρλο από το ΕΛΚΑ, τον Τίλης από το Ρινιού, τον Γκάντς από το ΙΣΙΕΡΕ, του Φρασίς, τον Δημήτρη από την ΚΟΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν αυτή τη φορά δείχνει ότι μπορεί να είναι ενωμένο και να προχωρήσει σε σημαντικά θέματα προς όφελος των πολιτών. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πνεύμα. Σίγουρα διαπραγματεύσει θα είναι δύσκολε μέχρι το Δεκέμβριο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Η συμφωνία αυτή των έξι πολιτικών ομάδων υπενθυμίσει τι προτεραιότητέ μα, τι κοινωνικέ συνέπειε, τι περιβαλλοντικέ, τι συνέπειε τη πανδημία, ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη δηλαδή όλε αυτέ. Θα πρέπει να βληθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας. Καμία χώρα από μόνη της δεν θα μπορέσει να τα καταφέρει. Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης περιορίζονται από το χρέος και μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορέσουμε να βρούμε νέους πόρους είτε μέσω κοινού χρέους όπως πρότειναν ο κύριος Μακρόν και η κυρία Μέρκελ ή με επιχορηγήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπαμε ότι δεν θα μπορέσει να συμφωνήσει με έναν πολιτές ε, πλαίσιο αν δεν υπάρχουν οι ίδιοι πόροι που ε, ζητούμε. Η κοινωνική κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Είμαστε στα τέλη του Μαΐου, έχουμε ήδη 25 βαθμούς, υπάρχει ξηρασία σε πολλές χώρες, πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες και πρέπει να αντέξουμε. Το περιβάλλον από την άλλη μεριά μπορεί να δημιουργήσει ε, 5 εκατομμύρια θέσει απασχόληση και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη μα. Έπειτα υπάρχει πολιτική συνοχή, η γεωργική πολιτική, τα κοινωνικά, ο πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η καταπολέμηση τη ανεργία. Θα το διαβάσετε το κείμενο. Πραγματικά αποτελεί καρπό εργασιών και έργου μα τρει μήνε. Είμαστε στα μέσα του δρόμου. Ο προπολογισμό του 2021 πρέπει να είναι στο ύψο που τον θέλουμε για να δώσει ελπίδα πρέπει η ελπίδα να καταστεί κάτι στο οποίο να μπορούν να προσβλέπουν οι άνθρωποι, όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι που ανησυχούν για το μέλλον τους και να μπορούν να πούν ότι ναι, η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος της. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριε Λαρουτούρ, κανονικά κύριε Χόλμαγερ τώρα στο σημείο 5 θα έπρεπε να πάρει το λόγο, αλλά με ενημέρωσαν ότι δεν έχει συνδεθεί ακόμα, οπότε πάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που είναι η ψηφοφορία για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για να χορηγήσει ενίσχυση στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, θα μιλήσω πορτογαλικά. Θα ήθελα από τη δικιά μου την πλευρά πάνω απ' όλα να επανέλθω στο θέμα των φυσικών καταστροφών. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι έκτακτη. Πάνω από 5 δισεκατομμύρια μπορέσαμε να κινητοποιήσουμε και εποφελούνται οι χώρες αυτές. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για 279 δισεκατομμύρια για την Ισπανία, την Ιταλία και την Αυστρία κυρίως. Η κινητοποίηση αυτή πρέπει να πούμε ότι γίνεται μέσω δανείων. Πρόκειται για μια αλληλεγγύη κυρίως με επιχορηγήσεις 100% και όχι με δάνεια διορθών, όχι με δάνεια. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε ότι η κινητοποίηση αυτή υπάρχει και αυτό φαίνεται και στην Πορτογαλία της Αζόρες για παράδειγμα, αλλά και ε, στην Ισπανία και στην Ιταλία και την Αυστρία που θα μπορούν να υποφεληθούν από αυτή την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, που είναι μια αλληλεγγύη που διαπιστώνουμε πολύ συγκεκριμένα στην πράξη. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να κάνω μια έκκληση να διατηρηθεί αυτό το Ταμείο. Να φροντίσουμε να υποφεληθούν πράγματι οι άκρος περιφερειακές περιοχές, γιατί αυτές είναι που αντιμετωπίζουν συνήθως προβλήματα από τις φυσικές καταστροφές. Και βέβαια οι εθνικές αρχές από τη δική τους την πλευρά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους πόρους αυτούς με όσο γίνεται περισσότερη διαφάνεια. Πρέπει να υπάρχει και μια αναλλαγικότητα ώστε τα αρνητικά να είναι όσο γίνεται λιγότερα. Μετά δηλαδή από τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Οι εθνικές αρχές δεν πρέπει να κρατούν τους σπόρους αυτούς για δικό τους όφελος, όχι, αλλά θα πρέπει να φροντίσουν αναλογικά, εξισορροπημένα, να βοηθήσουν αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο. Πρόκειται για ένα ταμείο αλληλεγγύης, μην το ξεχνάμε. Πρέπει να είναι λοιπόν ένα ταμείο το οποίο να κινητοποιεί πόρους γρήγορα, ώστε να είμαστε σε θέση να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι και αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, uh, Mr. Fernandez. Uh, I am Ευχαριστώ κύριε Φερνάνδε και μα ενημέρωσαν ότι η κυρία Χόλμαϊρ ακόμα δεν έχει συνδεθεί. Γι' αυτό θα περάσουμε από το σημείο 6 στο 7 για την πολιτική για τα κτίρια. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Κέλλερ, η οποία είναι μόνιμη εισηγήτρια για τα κτίρια και την κτηριακή πολιτική. Για να μα κάνει μια παρουσίαση. Five minutes, uh, Madame Keller. The floor is yours. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά, κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Πρόκειται για έγκριση της α, ε, ε, ε, έκθεσης για το κτίριο Βάη στο Στρασβούργο και θα σας παρουσιάσω μετά και τα συστήματα έγκρισης προειδοποίησης για δύο κτίρια στο Buenos Aires το ένα και ένα για την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, Εργασία στην ε, Πρατισλάβα. Και αν θέλετε, μπορώ να τα αναφέρω και τα τρία μαζί, κυρία, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε, ναι, βεβαίω. Για το ΒΑΙΣ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, το σχέδιο αυτό πρόκειται για ένα έργο ενίσχυσης της ασφάλειας του κτηρίου ΒΑΙΣ, εκεί που έχουμε και τις σημαίες το πρώτο σχέδιο λοιπόν εγκρίθηκε τον 28 Ιουνίου του 2018 για 11 εκατομμύρια ευρώ. Το σχέδιο αυτό είναι περίπλοκο και υπάρχουν ε, πολλά θέματα τα οποία μπλέκονται. Υπάρχουν διάφορε είσοδοι, την οποία ξέρετε και ε, για τους πεζού και για τα αυτοκίνητα. Και όπως ξέρετε, τίθεται το θέμα και τη ε, αισθητικής, προκειμένου να μην αλλάξουμε την αρχιτεκτονική του κτηρίου και να υπάρχει αρχιτεκτονική συνοχή και με το κτίριο Louis Weiss. Και σήμερα λοιπόν το έργο αυτό έχει φτάσει πλέον τα 27 εκατομμύρια ευρώ. Η είσοδος Louis Weiss, η οποία σήμερα γίνεται μέσα από προσωρινά κτίρια, παραπήγματα, για να γίνει ο επαρκετός έλεγχος ασφάλειας και να υπάρχει σωστή και ασφαλής πρόσβαση. Ε, γι' αυτό λοιπόν σας προτείνω να ψηφίσουμε υπέρ της έγκρισης ε, του, του έργου αυτού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύστημα έγκρισης προειδοποίησης, early warning, σε ό,τι αφορά ένα σχέδιο αγοράς κτηρίου για την αντιπροσωπεία στον Buenos Aires, το οποίο ήδη βρίσκεται ε, έχουμε προσωπία στον Buenos Aires. Θέλουμε λοιπόν να αγοράσουμε νέα γραφεία γιατί θεωρείται ότι τα παλιά, το, παλι, το παλιό κτίριο δεν είναι αρκετά ασφαλές. 14 εκατομμύρια ευρώ για 20 χρόνια, εκ των οποίων 8 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν στην αγορά για μια επιφάνεια 1.236 τετραγωνικών μέτρων για 24 άτομα. Θα υπάρχει και συμπληρωματικό εκμισθωτή για τρει υπαλλήλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την πνευματική ιδιοκτησία. Γι' αυτό λοιπόν σας προτείνω να μην εγκρίνουμε το ποσό που προβλέπετε για τις, τα, τις, ε, τα έργα, τα οποία μου φαίνονται δυσανάλογα σε σχέση με την ε, επιφάνεια. Τέλος, ε, η μελλοντική έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στην Βρατισλάβα για να τοποθετηθεί εκεί το, τα ιδρικά γραφεία της ΕΛΑ. Η κυβέρνηση της Σλοβακίας προτείνει να καταβάλει η ίδια το πόσο των 10 πρώτων ετών για την εγγύηση, για την ε, εκπίστωση. Στη συνέχεια θα επιφορτιστεί με το κόστος αυτός η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Εργασία που θα πρέπει να καταβάλει δηλαδή 1.020.000 για 5.500 τετραγωνικά μέτρα. Είναι ευαίσθητο λοιπόν το θέμα αυτό, γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε επί της ε, έντρας αυτής χωρίς να υπάρξει διαβούλευση και έτσι Διάφοροι σκιώδει συζητητέ εξέφρασαν την ανησυχία τους από αυτό και προτείνω στην υπηρεσία να ε, διαπραγματευτεί μία ρήτρα ευελιξία, λαμβάνοντα υπόψη και τη δυσκολία αυτή, που νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με την πόλη, αλλά μάλλον με τον τρόπο που αποφασίστηκε και εγκρίθηκε η πόλη αυτή. Αυτά λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αυτή είναι τα τρία θέματα που ήθελα να σας παρουσιάσω. Ευχαριστώ. πολύ, λέει ο πρόεδρος, προς την κυρία Κελέρ. Η κυρία Χολμαϊρ ακόμη δεν έχει συνδεθεί. Επομένω υπάρχει ο χρόνος. Έτσι δεν είναι. Έτσι υποθέτω. Ωραία. Οπότε έχουμε τον χρόνο, εάν θέλετε να ισχυώδες να λάβετε τον ε, λόγο. Εάν βεβαίως το επιθυμείτε. Οπότε πέστε μας, ε, είτε συνάντησή εδώ είναι αίθουσα, είτε από απόσταση, όχι από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει κανείς το λόγο. Καλά, τότε να περιμένουμε λίγα λεπτά την κυρία Χολμάιρ να συνδεθεί. Okay. Ως μικροφόνο, μιλά κάποιος στην αίθουσα. Ο πρόεδρος. Οπότε συνεχίζουμε στην ημέρηση διάταξη, ε, δηλαδή πάμε στην ε, ψηφοφορία να δούμε αν έχουμε απαρτία των 11 συναδέλφων που απαιτούνται για να γίνει ψηφοφορία. Οπότε παρακαλώ όλοι όσοι παρίστανται να πατήσουν το σχετικό κουμπάκι κάτω-κάτω στην ε, οθόνη της πλατφόρμας της Interactio. Τώρα γίνεται η καταμέτρηση. Since we have 13, we have reached... Είμαστε 13, επομένως έχουμε την απαρτία και με το παραπάνω, οπότε μπορούμε να κάνουμε εγκύρω στην ψηφοφορία. Σε αυτή την ψηφοφορία πρόκειται να ψηφίσουμε τις τροπολογίες που έχουν σχέση με τα εξή θέματα. Πρώτα πρώτα έχουμε την έκθεση όσον αφορά τι για ε, τη χρήση του 2021, τρίτο τμήμα του προπολογισμού. Δεύτερον, έχουμε το σχέδιο του προπολογισμού υπαριθμών 3 σε σχέση με το γενικό προπολογισμό του 20, ε, σε σχέση με το πλεόνασμα της χρήσης του 2019 και επίσης έχουμε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης προς ε, αρρωγή Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και Αυστρίας. Επίσης έχουμε μία και μόνη ψηφοφορία όσον αφορά την πολιτική ε, ακινήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κτίριο Λουίς Βάις ή στο Στρασβούργο. Έναρξη της ψηφοφορίας. And combination, declaring the vote open but immediately also suspending the ε, παραδόξως κήρυξα την έναρξη τη ψηφοφορίας αλλά τη λήξη της ε, συνεδρίασης. Οπότε θα τα ξαναπούμε στι 5 και μισή. Θα είναι και ο Επίτροπος ε, Χαν, ο οποίο θα μα παρουσιάσει τι αναθεωρημένες προτάσει τη Κομισιόν όσον αφορά του ίδιου πόρου, το πολιτισμό πλαίσιο, αλλά και τις ε, προτάσει για το σχέδιο ανάκαμψη και ανασυγκρότηση. Αύριο στι 4 η ώρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτή τη ψηφοφορία. Όμω έχουν ζητήσει οι δύο συνάδελφοι το λόγο ο κύριος Παπαδημούλης και ο κύριος Λεβαντόφσκι. Κύριε Λεβαντόφσκι, έχετε το λόγο. ευχαριστώ. Θέλω να σας πω ότι ψήφισα Yes, I am in voting. Ότι ψήφισα, ότι ψήφισα, λέγει ο κύριο Λεβαντόφσκι. Καλώς, καλώς, ελήφθη υπόψη. This closes our meeting for... Ωραία, εντάξει, τότε ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας ε, συνάντηση. Ευχαριστώ.